Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξη είναι η δήλωση του Συμβουλίου για την νομική βάση του μηχανισμού αξιολόγησης της Συμφωνίας του Σέγγεν. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία οφθαλμοσύλληψης catch the eye κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Kollege